ώστε να εδραιώσουμε περισσότερο και να κάνουμε πιο έντονη την πολιτική του Διεθνούς Οικοστηρίου σε συνεργασία από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, Επίτροπε. Έλεξε η συζήτηση αυτή. Η ψηφορία θα λάβει χώρα αύριο το μεσημέρι. Περνάμε τώρα στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης. Έκθεση ΛΙΣΕΚ σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για τη Συμφωνία Σύνδεσης ΕΕ Γεωργίας. Δίνω το λόγο στον εισηγητή τον κύριο και για τέσσερα λεπτά. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, κυρίες και κύριοι. Η έκθεση αυτή η έκθεση αυτή μεταξύ πολλών άλλων εκθέσεων που έχουμε εγκρίνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι πάρα πολύ σημαντική. Πολύ σημαντική και για μας, για τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίω όμως για την γεωργία και το κράτος και το λαό της χώρας αυτής που δίνουν πολύ μεγάλη σημασία στην έκθεση και στο μέλλον της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ίσως ως μέλος κάποια στιγμή. Υπάρχει και μια έκθεση η οποία αφορά τη Συμφωνία Σύνδεσης Ευρωπαϊκής Ένωσης Γεωργίας και τις διαπραγματεύσεις για τη σύναψη αυτής της συμφωνίας. Η έκθεση αυτή την οποία σας προτείνω, έχει να αντιμετωπίσει κάποια θέματα πάρα πολύ δύσκολα και λεπτά, τα οποία σχετίζονται με τη λειτουργία σήμερα του Γεωργιανού κράτους και με τις επιπτώσεις της σύγκρουσης του 2008, της σύγκρουσης με τη Ρωσική Ομοσπονδία. Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος που η έκθεση αυτή, έτσι όπως έχει συνταχθεί, με τη μορφή που έχει, έχει τύχη της μεγάλης υποστήριξης στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και ελπίζω να εγκριθεί ακριβώς από την παρούσα αρχική της μορφή. 35 ψήφοι υπέρ και μία αποχή. Αυτό ήταν το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας. Αυτό σημαίνει ότι όλες σχεδόν οι βασικές πολιτικές δυνάμεις ενέκριναν την έκθεση στην παρούσα της μορφή. Είναι μια έκθεση που στα μέσα ενημέρωσης ε, αποκαλείται πάρα πολύ θαραλέα. Και αν μπορώ να μιλήσω για λογαριασμό της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, η έκθεση αυτή μιλάει πάρα πολύ ξεκάθαρα και ντόμπρα για ζητήματα πολύ σημαντικά τα οποία έχουν να κάνουν ε, και με την Απχαζία και την Νότια Οσετία. Τι επαρχίε που έχουν αναγνωριστεί ω ανεξάρτητα κράτη από τη Ρωσική Ομοσπονδία. Κατά την άποψή μα όμω, και ελπίζω το ίδιο να πιστεύει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θα το δούμε μετά την ψηφοφορία. Ελπίζουμε, λέω, να κληθεί η Ρωσική Ομοσπονδία να σεβαστεί το διεθνέ δίκαιο. Πιστεύουμε ότι η κατάσταση όπου χιλιάδες ε, ε, άνθρωποι, χιλιάδες στρατιώτες, ρωσικά ε, στρατεύματα παραβιάζοντας και τις συμφωνίες που περάσαν το 2008 μεταξύ Γεωργίας και Ρωσίας που τις πρόθεσε ο πρόεδρος Σαρκοζή εκπροσωπώντας τότε την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να πάψει η παρουσία αυτών των στρατευμάτων. Και νομίζουμε ότι όλα αυτά τα γεγονότα w dokumencie e, Όλα αυτά τα γεγονότα λοιπόν εμείς τα αντιμετωπίζουμε ως κατοχή. Αυτό το λέμε σε όλα τα έγγραφα. Η παρουσία των στρατευμάτων στην Απχαζία και την Νότια Οσετία είναι κατοχή κατά την άποψή μας. Οι δύο αυτές επαρχίες αποτελούν ένα απόσπαστο τμήμα της επικράτειας της Γεωργίας και είναι ένα κατεχόμενο έδαφος, ένα κατεχόμενο εδάφι. Και αυτό είναι το πολιτικό στοιχείο, αν θέλετε, αυτής της έκθεσης, αλλά υπάρχουν και άλλα, και άλλα στοιχεία η συμφωνία για την ε, Συμφωνία ελεύθερων, ε, για τη Ζώνη Ελεύθερων Συναλλαγών. Ε, δυστυχώς δεν έχω χρόνο για να αναφέρω όλα αυτά τα ζητήματα. Σας ευχαριστούμε, λέει Πρόεδρος. Έχουν αρκετοί ζητήσει το λόγο στη δικασία Catch the Eye. Η κυρία Ντάντσι λένε πρώτη. Πολύ σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζει τις προσπάθειες της Γεωργίας όσον αφορά τις κοινέ αρχές και αξίες της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου, των δικαιωμάτων του ανθρώπου στην πολιτική καλής γειτονίας αλλά και μέσω της κοινοβουλευτικής διάστασης όσον αφορά την ανατολική εταιρική σχέση προς τα κράτη της Ανατολικής Ευρώπης και όσον αφορά και την ευρωμεσογειακή ε, κοινοβουλευτική διάσταση. Ελπίζουμε ότι οι αρχές στη Γεωργία θα καταβάλουν κάθε προσπάθεια, θα κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους, ώστε να δημιουργηθεί ένα θετικό κλίμα όσον αφορά την προσέγγιση των ε, ευρωπαϊκών προδιαγραφών όσον αφορά την κατάρτιση, εκπαίδευση, την ε, θετική ε, ένταξη των εθνοτικών μειονοτήτων αλλά και της πολιτικής γειτονίας. Με ένα θετικό επικοδομητικό διάλογο και με τους εκπροσώπους της αντιπολίτευσης. Η αντιπολίτευση πρέπει χωρίς προσκόμματα να έχει πρόσβαση στα μέσα ενημέρωσης. Η Γεωργία πρέπει να είναι εταίρος μας. Πρέπει να προσεγγίσει περισσότερο την Ευρωπαϊκή Ένωση αυτός ο εταίρος μας, η Γεωργία. Και γι' αυτό απαιτείται οι πολίτες να έχουν διευκολυμένη ε, πρόσβαση σε θεωρήσεις διαβατηρίων ώστε να ταξιδεύουν ευκολότερα προς την Ευρώπη. Σας ευχαριστώ και εγώ Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω τον συνάδελφο για την σύνταξη αυτής της έκθεσης, τον συνάδελφο Ντίσεκ. Η Γεωργία έχει σημειώσει πρόοδους όσον αφορά τις ε, δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις. Η συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι θετική ευρωπαϊκή δράση. Υποστηρίζουμε την ευρωπαϊκή προοπτική της γεωργίας. Όσον αφορά την διατήρηση της προώθησης των διαπραγματεύσεων για την σύνδεση, καθώς επίσης και για τις διαβουλεύσεις και διαπραγματεύσεις για μια διευρυμένη ζώνη συναλλαγών. Είναι σημαντικό να εμπλακεί η Ευρωπαϊκή Ένωση στην επίλυση των θεμάτων σύραξης και των τριβών όσον αφορά τις νέες ευθύνες που πρέπει να επομισθούν όλοι σε σχέση με την πολιτική γειτονία. Χαιρετίζουμε και τη διεύρυνση της εντολή όσον αφορά αυτέ τι διαβουλεύσει και το διευρυμένο πλαίσιο. Πρέπει να διασφαλιστούν οι προποθέσει ε, για τις ε, κατεχόμενες περιοχές. Πρέπει επίσης η συμφωνία μεταξύ Γεωργίας και Ρωσίας ε, να ληφθεί υπόψη όσον αφορά την ένταξη της Ρωσίας στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου. Ελπίζουμε ότι νέες οδοί για την σταθεροποίηση της περιφέρειας αυτή θα εξευρεθούν. Ναι, ε, νομίζω ότι η δημιουργία και η πρόθεση της ε, δημοκρατίας ήταν από τα πιο δύσκολα θέματα που άφησε παρακαταθήκη η πρώην Ένωση Σοβιετικών Δημοκρατιών. Για τη Γεωργία συγκεκριμένα είχαμε διάφορα προβλήματα και ιδιαίτερα το θέμα της Απχαζίας ε, ως ε, θέμα ακαθόδες μοιάζει πολύ με το κοσυφοπαίδιο. Βεβαίως η δημοκρατία στην Γεωργία χρειάζεται την προσοχή μας, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο η επιρροή μας στην ε, περιοχή επαρκεί. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τέλος η κυρία Λούνατσεκ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Λίσεκ για την πολύ καλή έκθεση και την πολύ καλή συνεργασία με τις διάφορες ομάδες και εμείς στους πράσινους την υποστήριξαν την έκθεση αυτή στην Επιτροπή και θα το κάνουμε και αύριο. Να τονίσω όμως ένα θέμα που είναι σημαντικό γιατί όσο και αν επέκρινα τη Ρωσία για την κατοχή εδαφών της Γεωργίας παρόλα αυτά θα πρέπει να δούμε ακριβώς τι συνέβη το 2008 έχουμε τροπολογίες που θα θέλαμε να περιληφθούν στην έκθεση και νομίζω επίσης θα πρέπει η Γεωργία να συνεργαστεί περισσότερο με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Έχουμε και την ε, Επιτροπή Νορβηγική του Ελσίνκη που λέει κάθαρα και την έκθεση της που λέει κάθαρα ότι οι αρχές Γεωργίας θα έπρεπε να είχαν προσέξει ιδιαίτερα τι είχε συμβεί μετά από τις πανικές δραστηριότητες του 2008 και ότι και τα δύο μέρη δεν είχαν την διάθεση να συνεργαστούν και να διεξάγουν τις απαραίτητες έρευνες μετά από τη σύραξη του 2008. Λένε και εφημερίδες στην Γεωργία ότι ο πρόεδρος Σάκασφίλη άφησε τους Ρώσους να τον προκαλέσουν και προκάλεσε ρήγματα στο ΝΑΤΟ. Δεν ξέρω ακριβώς λοιπόν τι συνέβη, αλλά ό,τι και να έχει συμβεί θα πρέπει και η ΟΗΕ να συνεργαστεί όσον αφορά την, κατα... την καταπάτηση ανθρωπινών δικαιωμάτων. Ευχαριστώ. Επίτροπε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Κοινοβούλιο για την δέσμευσή του όσον αφορά την συμμετοχή στις διαπραγματεύσει με την Γεωργία. Είχαμε πολύ καλή εργασία από τους ηγητές που μας βοήθησαν να προετοιμάσουμε μια ισορροπημένη έκθεση. Οι συστάσεις αυτής της έκθεσης ήταν πάρα, πολλές, πάρα πολύ χρήσιμες στις περιπτώσει ε, διαπραγματεύσεις με την Γεωργία. Διαπραγματεύσεις που θα πρέπει να έχουν ως τελικό αποτελέσμα την ενσωμάτωση της Γεωργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζουμε την σημασία προς τη γεωργία στην ευρωπαϊκή της ταυτότητα και οποιαδήποτε όμως αναφορά στο άρθρο 49 παραμένει επίμαχη για τις χώρες μέλη και θα πρέπει να λυθεί το θέμα αυτό. Είναι σημαντικό για τη γεωργία αυτή τη στιγμή να υποφεληθεί στο μέγιστο των πολιτικών ευκαιριών που της παρέχει η πολιτική σύνδεση και η πολιτική ολοκλήρωση τη στιγμή αυτή ώστε να δημιουργηθεί περισσότερη Ευρώπη στο εσωτερικό τη Γεωργία. Χρησιμοποιώντα λοιπόν αυτή την ευκαιρία, θα ήθελα να σα ενημερώσω για την κατάσταση των διαπραγματεύσεων με του Γεωργιανά, με τους Γεωργιανούς ε, συναδέλφους μας έχουμε επαφές και ξεκινήσαμε από τον Ιούλιο 2010 επαφές σε γενικές συνελεύσεις καλύπτοντας διάφορα θέματα ασφάλεια, δικαιοσύνη οικονομική συνεργασία και είχαμε 7 συνελεύσεις ολομελίας που έχουν λάβει χώρα μέχρι στιγμής Έχουμε συζητήσει του γενική, τους αρχέ τη αρχές της συμφωνίας και προσωρινά συμφωνήσαμε επί ενός, Εβραίου, ενός ε, μεγάλου κειμένου ώστε να ενισχύσουμε το διάλογο για την ασφάλεια. Και βεβαίως η ασφάλεια και η ειρήνη μετά από τις διάφορες ε, συγκρούσεις που είχαμε στην περιοχή αποτελούν από τα πιο σημαντικά θέματα για τους Γεωργιανούς και οι δύο πλευρέ προχώρησαν και πρόοδευσαν όσον αφορά την οικονομική συνεργασία. 19 κεφάλαια έκλεισαν προσωρινά σε σύνολο 28. Δεσμεύτηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση να ξεκινήσει, να ξεκινήσει διαπραγματεύσει με την Γεωργία ώστε να συνταχθεί το ταχύτερο δυνατόν η μελλοντική συμφωνία σύνδεση. Είχαμε και διάσκεψη κορυφή στην Βασοβία 29.30 και θα πρέπει να πιέσουμε την Γεωργία ώστε να εφαρμόσει κάποιες σημαντικές συστάσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση κατανοεί τις προσπάθειες που έχει κάνει η Γεωργία για την πρόοδο των διαπραγματεύσεων. Βρισκόμαστε τώρα στα τελικά στάδια των διαπραγματεύσεων και μέχρι το τέλο η Κομισιόν θα είναι σε θέση να υποβάλει την επίσημή τη σύσταση προ χώρε μέλη. Μάλιστα, να τονίσω ότι έχουμε και μια σημαντική ε, συμφωνία μεταξύ Γεωργίας Ρωσίας για την προσχώρηση της Ρωσίας στον Παγκοσμίο Οργανισμό Εμπορίου. Καλωσορίζουμε και το συμβασμό που, και συμβαστική λύση που, βρήκε η Γεωργία με τη Ρωσία για πρόσβαση στον Παγκοσμίο Οργανισμό Εμπορίου και η κυρία Άστον επισκέφθεται σήμερα τη Γεωργία και θα έχει επαφές με τον πρόεδρο Σακασφίλη με κύριο στόχο να ενισχύσει το μήνυμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την συνεχή της δέσμευση με τη Γεωργία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 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι